Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ακρόαση με τον υποψήφιο Επίτροπο για την Πολιτική Γειτονίας και Διεύρυνσης, και καλωσορίζω τον Ιωάννης Χάν. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που περνάτε την διαδικασία, ήσασταν επίτροπος ήδη για τα περιφερειακά και κάποια από τα πράγματα που σας απασχολούσαν εκεί, δηλαδή η ανοικοδόμηση κάποιων περιφερειών, είναι επίσης ε, στη δουλειά και του νέου σας χαρτοφυλακίου με μια επιπλέον δυσκολία. Θα πούμε πρώτα απ' όλα κάποια τεχνικά ζητήματα. Ο υποψήφιος επίτροπος ε, μπορεί να μιλήσει, θα βγάλει μια ομιλία για 15 λεπτά. Μετά θα γίνουν οι ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση θα κρατήσει ένα λεπτό και θα έχει ο υποψήφιος 1,5 λεπτό στη διάθεσή του για να απαντήσει. Μετά μπορεί σε 30 δευτερόλεπτα να τεθεί μια συμπληρωματική ερώτηση και απάντηση μετά σε ένα λεπτό. Οι συντονιστές ε, θα έχουν μια πιο προνομιακή μεταχείριση σύμφωνα με τη συμφωνία που κάναμε. Θα έχουν 4 λεπτά δηλαδή αντί για τρία λεπτά για τις ερωταποκρίσεις και επειδή είμαστε και ευγενικοί το ίδιο θα γίνει και με τον Μπέρντ Λάγκε πρόεδρο της Επιτροπής ΙΝΤΕ. Κανονικά έπρεπε να έχει τρία λεπτά οπότε εμείς είμαστε γενναιόδοροι και του δώσαμε τέσσερα και μετά τους συντονιστές και τους δύο προέδρους ε, των ε, δύο ε, που επιτροπών θα περάσουμε στον κανονικό ρυθμό. Μετά θα μπορέσουν οι ομάδες όπως είπα να θέσουν ερωτήσεις ομαδών αλλά οπωσδήποτε και οι μικρότερες ομάδες θα μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους. Θα σας πω μόνο το εξής. Εγώ παρακολούθησα και χτες ακρόαση. Θα είμαι αμήλικτος. Θα κόβω μικρόφωνα. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε με τις ερωτήσεις. Αν χάσουμε το ρυθμό βεβαίως αδικούμε και τους συναδέλφους που είναι τελευταίοι στον κατάλογο. θα χρονομετράει η γραμματεία και όταν τελειώσει ο χρόνος τελείωσε. Τα γνωστά δηλαδή, όχι κύριε πρόεδρε, τελευταία μου παρατήρηση και τα λοιπά, δεν θα περάσουν. Και ζητάω την κατανόησή σας για την διαδικασία. Θεωρώ πως ο κύριος Χάν έχει ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο. Αν δούμε τις εξελίξεις ε, στην ανατολική γειτονιά μας ε, βλέπουμε πως είναι περίπλοκα τα πράγματα. Στην νότια γειτονιά μας οι γειτονές μας είναι γείτονες της Ευρώπης ε, και εκεί πέρα ε, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη για να μην πω ότι είναι δραματική. Και σε αυτό το περιβάλλον θα αναλάβει καθηκόντα ο κύριος Χάν. η Επιτροπή Γιούγκερ θα συνεχίσει να εργάζεται για την διεύρυνση, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθούν σε αυτή την περίοδο οι διαπραγματεύσεις. Οπότε, ε, σημαίνει αυτό κύριε Χάν πως εξακολουθούν να υφίστανται οι υποχρεώσεις μας απέναντι στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Και επίσης ε, για την διαπραγματευτική εντολή για την Τουρκία ισχύει αυτό το οποίο αναφέρεται στην εντολή ότι τελικός στόχος είναι η ένταξη. Παρά το ότι υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στις διαπραγματεύσεις. Και έχουμε άρα αυτές τις ανοιχτές διαδικασίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μας αναπτύξετε κάποιες πρώτες σκέψεις για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχετε